Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll θα επανάληψη τη Συνόδου. Τα πρακτικά της, χθεσινή συνεδρίαση τα έχετε στη διαθεσή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ενστάσει. Όχι, μάλιστα. Άρα τα πρακτικά εγκρίνονται. Από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και την... Ε, έλαβα επίση και την ε, τοποθέτηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.